είχαμε φτάσει σε αυτή την επιτυχία και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε συνεισφέρει υπέρ του ευρωπαϊκού κοινού, των επιχειρήσεων και της κοινότητας. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα παρακαλέσω και εσάς και τον Επίτροπο κύριο Ρέν, αλλά και την εισηγήτρια να προχωρήσετε στο τραπέζι που έχουμε βάλει στο κέντρο της αίθουσας ώστε να μπορέσω και εγώ να κατέλθω και να συνυπογράψουμε όλοι το κείμενο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πρακτικά της χθεσινής συνεδριάσεως έχουν ήδη διανεμηθεί. Παρακαλώ, έχετε ενστάσεις. Όχι. Καλώς. Θεωρώ ότι εγκρίνονται τότε τα πρακτικά αυτά. Σύμφωνα με την ημερησία διάταξη, ακολουθεί δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για τα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής G20. Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, στις 2 Απριλίου 2009 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 20 χωρών συνήλθαν στο Λονδίνο για να συζητήσουν